Λαμπάγιοβα, κοινή επιχείρηση Shift to Rail. Α, αποφασίζουμε για την απαλλαγή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύλλογο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ για τα λουλούδια.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 Κυρίες και κύριοι, ο Πρόεδρος. Κύριε Λίντς, κύριε Λίντς, παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν έχουμε ψηφορίες για των γνωμοδοτήσεων της ΕΝΒΗ σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό θα ισχύσει και ε, ρωτώ την παρακαλώ ε, όσοι δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη συζήτηση να αποχωρήσουν Ή κάντε ησυχία ή παρακαλώ βγείτε από την αίθουσα. Και μπείτε. σας παρακαλώ. Πολύ ωραία. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έκθεση Ντάλι. Πρώτη επιδόσεων η τι εκπομπέ από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Πρώτο ομιλητή, συγγήτρια, κύριε Ντάλη. Παρακαλώ. Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές με τους οποίους συνεργάστηκα. Ευχαριστώ για το όραμα, ευχαριστώ για τις απόψεις, τις ιδέες που καταθέσατε που με βοήθησαν να διατυπώσω την τελική μας πιο φιλόδοξη θέση. Εργαστήκαμε σκληρά, είχαμε επίπονες διαπραγματεύσει όμως σήμερα είμαστε εδώ γιατί η συναντήληψη είναι πλέον ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος, μπορούμε να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων και να κάνουμε τις χώρες μας πιο ανταγωνιστικές. Η νομοθεσία για εκπομπές των λόγω οχημάτων είναι μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης που ζητά να περάσουμε από παλαιότερα πρότυπα σε νέες τεχνολογίες σε έναν χώρο καινοτομία, σε έναν χώρο όπου οι επενδύσεις πηγαίνουν στην έρευνα και την καινοτομία. Οι στόχοι μείωση των εκπομπών συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου για το 2025 και το 2030. Όμως αυτά είναι η αρχή και μόνο στην πορεία προς την οικονομία του μέλλοντος. Μετά από σειρά συναντήσεων με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατορθώσαμε να συναπολογίσουμε το 37,5 μείον στις εκπομπές για τα επιβατικά αυτοκίνητα και 31 για τα φορτηγά. Τα μη φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα θα εκπέμπουν ακόμη λιγότερο στο μέλλον. Οι κυψέλες υδρογόνου, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όλα αυτά θα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή και χαίρομαι που προς εκεί πηγαίνουμε. Ο δεν ήταν εύκολος, αντιμετωπίσαμε δυνατά λόμπι και τις αντιδράσεις και κάποιων κατών Αλλά τι είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή. Καταφέραμε παρόλα αυτά να κλείσουμε κάποια παραθυράκια τα οποία θα είχαν αποδυναμώσει την εν λόγω νομοθεσία. Οι κατασκευαστές εν ώψη των νέων κύκλων ε, μέτρηση εκπομπών δεν θα μπορέσουν να παρουσιάσουν τεχνητά βελτιωμένα αποτελέσματα. Μέσω αυτού του νέου μηχανισμού λοιπόν θα μειώσουμε τις εκπομπές και στο δρόμο, όχι μόνο στο εργαστήριο. Αναγνωρίζουμε την σημασία των νέων υποδομών. Εν προκειμένου υιοθετήθηκε η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρέχουμε ε, περισσότερες υποδομές σε περισσότερα σημεία σε όλη την Ευρώπη, κατά το οποίο θα πετύσει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Κατανοώ βεβαίω τις ανησυχίες των συνδικάτων. Στο πλαίσιο αυτό επιβαρύνουμε με ε, τίμημα τις ε, υπερβολικές εκπομπές έτσι ώστε να μην υπάρξουν και υπερβολικά δυσμενεί κοινωνικέ επιπτώσει. Για να τονώσουμε επίση και την απασχόληση, λάβαμε μέτρα κάτι το οποίο είναι προτεραιότητα και για μένα. Η νέα νομοθεσία σημαίνει εξοικονόμηση στα καύσιμα και πιο φτηνά, πιο προσιτά τα χαμηλών μηδενικών εκπομπών. Πιστεύω ότι πρόκειται για τη σωστή κατεύθυνση η πολιτική πρέπει να προχωρήσει προς πιο καθαρές μεταφορές και εμείς ως πολιτικοί πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτήν την κίνηση και να τονώσουμε βεβαίω και τη ζήτηση όπως θα γίνει πιστεύω με την ελόγω νομοθεσία. Έτσι θα τονώσουμε και τη βιομηχανία μας, θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις που απαιτούν δεξιότητες και θα τονώσουμε την οικονομία μας που εκπροσωπεί το 4,2% της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ τους πάντες για τη συνεισφορά τους, ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές και κάθε άλλον που συνεργάστηκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγος των Επίτροπο Αρίας Κανιέτη. Παρακαλώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, θα ήθελα να φτάσουμε σε ε, ένα συμπέρασμα για την περίοδο μετά το 2020 για τα ελαφρά οχήματα. Πρόκειται για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα για τα βαρέα οχήματα, έτσι ώστε να έχουμε καθαρή ενέργεια μέχρι το 2030. Ε, μέσα στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης των δύο θεσμικών οργάνων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νταλή για την ηγετική της ε, θέση. Αυτό σήμανε πολύ μεγάλη και ουσιαστική εργασία για να είναι επικεφαλή των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους Σκιώδης. Η συμφωνία είναι φιλόδοξη και ισορροπημένη, έτσι ώστε να ρυθμίσουμε τις εκπομπές ε, διοξίδιου του άνθρακα. Ο, ο στόλος ε, των αυτοκινήτων θα πρέπει να προβεί σε μία μείωση ε, κατανάλωσης ε, καυσίμων, μάλλον μείωση ρήπων της τάξης του 37,5% και 31% μετά το 2030. Χρειάζεται ένα ε, καινοτόμο ουδέτερο σύστημα έτσι ώστε να έχουμε μηδενικές εκπομπές και ένα σύστημα χρηστής διακυβέρνησης έτσι ώστε να έχουμε μείωση εκπομπών όχι μόνο σε επίπεδο εργαστηρίου. Μία αναθεώρηση θα γίνει το 2023, έτσι ώστε ο τομέας των μεταφορών θα κινηθεί προς την καθαρή κινητικότητα. Θα ήθελα να μιλήσω για τα ευεργετήματα. Ε, τα συμπεράσματα αυτά θα φτάσουν σε μείωση εκπομπών κατά 24% μέχρι το 2030. Αυτό αφορά τα βαρέα οχήματα ιδιαίτερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανταποκριθεί στη Συμφωνία του Παρισιού έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν καθαρότερο αέρα και οι καταναλωτές να ευεργετηθούν ε, και οικονομικά, δηλαδή θα εξοικονομήσουν 1.100 ευρώ μέχρι το 2030 και αυτό μέχρι 4.000 συνολικά. Έτσι θα εξυγχρονίσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία και θα προωθήσουμε την καθαρή τεχνολογία. Το σύστημα κινήτρων για μηδενικές εκπομπές θα οδηγήσει σε μία νομοθεσία έτσι ώστε να έχουμε 35 εκατομμύρια οχήματα χαμηλών εκπομπών. Ο νέος κανονισμός θα έχει και θετικό αντίκτυπο ε, οδηγώντας σε 60.000 νέες θέσεις εργασίας. Η ε, Συμμαχία των Συσσωρευτών δημιουργήθηκε για να δημιουργήσουμε μία σωστή αλυσίδα και νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, ε, φτάνουμε σε μία μετάβαση μηδενικών εκπομπών το 2030 το 87% των οχημάτων θα έχουν μία, ακόμα μία μηχανή εσωτερικής καύσης σε σχέση με τα υβριδικά. Όμως θα γίνουν οι κατάλληλες επενδύσεις και ε, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Αυτό αφορά και τη διαδικασία αναμετάδοσης. 2,5 εκατομμύρια σημεία ε, ανατροφοδότησης θα υπάρχουν στους δρόμους για τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αγαπητά μέλη, θα ήθελα να υποστηρίξετε αυτή τη φιλόδοξη συμφωνία που θα ψηφιστεί αύριο. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχει εκδώσει μία ανακοίνωση η Επιτροπή για να υποστηρίξουμε την συνολική συμφωνία, έτσι ώστε η Ευρώπη να μεταβεί στην καθαρή κινητικότητα και σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ντέλη από την Επιτροπή Μεταφορών. Κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ πρόκειται για αστείο. Ο πρόεδρος του λόμπι των Κρασκευαστών, ο κύριος Ταβάρες, μας προσέβαλε εμάς, το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό σώμα. Μα είπε ότι είμαστε ερασιτέχνε, γιατί θέλουμε, λέει, να μειώσουμε τι εκπομπέ των αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Ερασιτέχνε, λέει, γιατί αφού γκραζόμαστε του νέου που διαδηλώνουν για το κλίμα. Ερασιτέχνε, γιατί κάνουμε αυτό που ε, υπαγορεύει η αίσθηση ευθύνη. Ναι, να μειώσουμε τι εκπομπέ που οφείλονται στι οδικέ μεταφορέ. 37,5% μείωση για τα ελαφρά οχήματα. Όχι αύριο, για το 2030. Αυτοί οι οποίοι αναβάλουν τη μάχη για το κλίμα είναι οι σκεπτικιστές, αλλά που δεν βρίσκονται δυστυχώς για αυτούς στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε το συντομότερο δυνατόν τις εκπομπές, γιατί είναι καλό για το κλίμα και είναι καλό και για την απασχόληση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος το Παρακαλώ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, για την ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Αύριο θα ε, ψηφίσουμε πολύ πιο αυστηρές τιμές για τις εκπομπές καυσαερίων από τα ελαφρά. Μέχρι το 2030 θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά πολύ οι εκπομπές και θεωρούν μάλιστα κάποιοι ότι είναι πολύ χαμηλές, άλλοι ότι είναι υπερβολικές οι οριακές τιμές που προτείνουμε. Εγώ να σας πω όμως ότι δεν θα είναι και παιχνιδάκι να πετύχουμε τις οριακές αυτές τιμές με τα αποτελέσματα ε, που είχαμε βελτιώσαμε τις προτάσεις ε, της Κομισιόν. Αν σκεφτεί κανείς τι ε, ξεκίνησε να συζητά εδώ το κοινοβούλιο. Θέλαν 50% στους 75% θέλαν οι πράσινοι και όλα αυτά ήταν παράλογα, μη ρεαλιστικά και ότι θα καταστρέφονταν και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Υποτίθεται ότι η ηλεκτροκίνηση θα έπαιρνε την πρωτοκαθετρία και θα είχαμε μηδενικές εκπομπές. Έχουμε όμως ρεαλιστικούς τώρα στόχους για το 2025, το 2030 θα επιβεβαιώσουμε, θα παληθεύσουμε πού βρισκόμαστε και θα δούμε αν μπορούμε και με το 31% για τα ελαφρά επαγγελματικά να ε, προχωρήσουμε. Σίγουρα θα θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στις καινοτόμες ε, τεχνολογίες ε, για κάποια καύσιμα. Για ιδεολογικούς λόγους δεν υπήρξε πλειοψηφία για τεχνολογικά ουδέτερες λύσεις και έτσι χάσαμε μια ευκαιρία. Εγώ πάντως θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την τεχνολογική ουδετερότητα. Πάντως αυτό το νομοθέτημα, αυτό το συμβιβασμό πρέπει να τον περάσουμε. Χρειάζεται να δώσουμε στους καταναλωτές και στους χρήστες ασφάλεια ε, μέχρι το 2025 να ξέρουμε τι πρόκειται να ε, υπάρξει για τα αυτοκίνητα. Ήδη έχει μπει σε κυκλοφορία το νέο σύστημα. κύριο κύριος Βέλκεν τώρα εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Αξιότιμε πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θέλω να πω και πάρα πολλά γιατί δεν έχουν προηγηθεί εντατικές συζητήσεις. Νομίζω ότι με αυτόν τον κανονισμό πράγματι ε, προχωρούμε προς μια κινητικότητα πιο καθαρή η οποία θα φροντίζει επίσης ε, και για να πληρώνουν λιγότερο οι καταναλωτές. Ε, είναι καλό. Έχουμε λοιπόν μια αλλαγή στον τομέα των μεταφορών και είναι καλό να συνδιαμορφώσουμε εμείς την κατάσταση βάζοντας το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις. Όσο σοσιαλδημοκράτες όμως έχουμε και ευθύνη απέναντι στους εργαζομένους. Εξού και είναι σημαντικό ο κανονισμός αυτός, αντίθετα με αυτό που είπε ο συνάδελφος ε, Γκίζικ, πρέπει ε, να ε, χαρακτηρίζεται από άνοιγμα τεχνολογικό. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα καύσιμα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που θέλουμε να τα αποκλείσουμε διότι πρόκειται για καύσιμα που μπορούν να καταναλώσουν, να καλύψουν πάρα πολύ πολύ μεγάλες εκτάσεις ε, και αυτό δεν είναι απόλυτα ε, παραγωγικό. Εμείς για το μέλλον αυτό που πρέπει να φροντίσουμε είναι η δίκαιη μετάβαση. Αυτό πρέπει να είναι στο επίκεντρο και θα πρέπει ε, να προωθήσουμε και την επιμόρφωση ε, με περισσότερη χρηματοδότηση, να κοιτάξουμε το μέλλον, ε, ε, για να λάβουμε υπόψη και το ωράριο το εργασιακό και την κατανομή της εργασίας. Είναι σημαντικές αυτές οι ευθύνες για τους νομοθέτες και με γνώμονα πάντα και την αλλαγή του κλίματος, έχοντας υπόψη και τις διαδηλώσεις των νέων που θέλουν να τους αφήσουμε έναν πλανήτη υγιή στο μέλλον. Ευχαριστώ. Πρώτος ευχαριστώ. Ε, μπλε κάρτα από τον κύριο Ρούμπικ την δέχεστε στα γερμανικά. Κύριος Ρούμπικ, ε, ε, θέλει να σας θέσει μια ερώτηση. Τη δέχεστε, όχι. Οι συνάδελφοι από τη Τσεντιού θα πρέπει να μάθουν να συμπεριφέρονται και όχι μετά να οριώνται και να σύουν τις μπλε κάρτες. Δεν αντιδεχτώ. Οπότε λέει ο Πρόεδρος. Συνάδελφοι, σήμερα ζήσαμε πολλέ διαφωνίε, αλλά δεν είναι όλο το θέμα. Οι φωνασκίες δεν είναι ευχάριστες. Λοιπόν, Mess Μάκερ από την ECR, παρακαλώ. Από την Κυριακή, Πρόεδρε, κάποιες δεκάδες ε, νεαρών στρατοπεδεύουν έξω από το Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ζητώντα την υπερψήφιση νόμου για το περιβάλλον στο Βέλγιο. Έχει μια συμβολική σημασία αυτό. Ήρθε καιρό για δράση. Θέσαμε στόχου, ας κοιτάξουμε να τους πετύχουμε. Υπάρχει στη Φλάνδρα ένα σχετικό σχέδιο νόμου. Λοιπόν, ας κάνουμε αυτό που πρέπει και εμείς. Έχουμε μπροστά μας ένα φιλόδοξο πακέτο που αποτελεί το πράσινο φως για φιλόδοξα μέτρα. Το 37,5% βέβαιος, λιγότερες εκπομπές. Το NBA, το κόμμα μου στη Φλάνδρα, υποστηρίζει αυτή την κίνηση. Στο Βέλγιο η αντίστοιχη μείωση είναι 25%. Χρειαζόμαστε λοιπόν καινοτόμε τεχνολογίε για να μειώσουμε τι εκπομπέ στην πηγή και να πετύχουμε του στόχου για την προστασία του περιβάλλοντο. Επίση, Θέλουμε πρασίνισμα του στόλου των αυτοκινήτων, θέλουμε καλύτερη τεχνολογία. Αυτό θα προσελκύσει επενδύσεις στην καινοτομία και στην ποιότητα στις πόλεις μας και στα χωριά μας. Οι πόλεις μας δικαιούνται καθαρό αέρα. Αν η Ευρώπη φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί την Κίνα, πρέπει οι κατασκευαστέ μας να καινοτομήσουν και να αρχίσουν να παράγουν οχήματα χαμηλότερων εκπομπών. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε και όχι σε λογισμικό το οποίο διευκολύνει του απαταιώνε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριο Τόρβαλς, εκ μέρου των φιλελευθερών Τσαλντε. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Να πω πρώτα κάποια καλά λόγια για την Μυρία Μιτάλη, γιατί όπως μάλλον γνωρίζετε, πέρασαμε λίγο δύσκολα με το Συμβούλιο χωρίς την Μίριαμ και την επιμονή της, το αποτέλεσμα φοβούμαι θα ήταν πολύ διαφορετικό. Μίριαμ, ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Λοιπόν, λίγες γενικές πληροφορίες χρειάστηκε, να τα βάλουμε όλα κάτω. Στην Φιλανδία, ένα αυτοκίνητο θα εξέπεμπε 48 γραμμάρια ένα χιλιόμετρο. Γιατί, γιατί το μείγμα στο οποίο βασίζεται η παραγωγή ενέργειας είναι διαφορετικό. Στη Γερμανία οι εκπομπέ ήταν 131 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο λόγω του τρόπου παραγωγή τη ενέργειας. Και γι' αυτό το λόγο δυσκολευτήκαμε, διότι στη μέση τη νύχτα περιμένουμε τηλεφώνημα από το Βερολίνο. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώ. Το θέμα είναι ποιο είναι το μείγμα παραγωγή ενέργεια το οποίο παίρνουμε δεδομένο. Εάν δεν γίνει εκεί προσπάθεια, τότε θα αποτύχουμε όλοι μας. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο. Αυτό είναι ένα γεγονός. Διότι το παλιό μου ντίζελ που είναι 7 ετών με το βιοκαύσιμο παράγει λιγότερο διοξίδιο σε σύγκριση με ένα ηλεκτρικό όχημα στη Γερμανία. Οπότε αγαπητοί φίλοι οι Γερμανοί προσπαθήστε κάτι πρέπει να κάνετε Πρέπει να βελτιώσετε την τεχνολογία σας και αλλάξτε. Αλλάξτε. Αν δεν αλλάξει ο τρόπος παραγωγής ενέργειας και το σχετικό μείγμα, τότε εσείς θα χάσετε. Ευχαριστώ. σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έκχουτ από τους πράσινους ένα μισή λεπτό. Έχουμε μια ε, μπλε κάρτα, την δέχεστε. Κύριε Τόρβαλτς, Θέλω να ρωτήσω, λέει ο κύριος Λίζα, τον κύριο Τόρβαλτσα, αν έχει καταλάβει ότι στο ETS έχει ανέβει από πάνω από 20 ευρώ η τιμή ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ε, και επειδή φεύγουμε από τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια στη Γερμανία και από ε, αυτή τη μορφή ενέργειας χρήση του άνθρακα, ε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς ε, να το παραγνωρίσει. Ευχαριστώ. Με μεγάλη ικανοποίηση να απαντήσω, λέει ο κύριος Τόρβαλ, στα γερμανικά. Έχω διαβάσει όλες τις εκθέσεις της Επιτροπής για του Άνθρακα για τη, από τη Γερμανία. Για το 36 γίνεται λόγος εδώ, έτσι, αν έχω διαβάσει καλά, για το 2036. Άρα, για να καταφέρουμε κάτι, χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη ταχύτητα. Ευχαριστώ λοιπόν. Συνεχίστε με μεγάλη ενέργεια και ενεργητικότητα για να τα αλλάξουμε όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς. Ε, ο κύριος, Φαν... τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Μίρια Μντάλη για την εξαιρετική εργασία. Δώσαμε μεγάλη μάχη και είχαμε πολλές διαφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλοί δεν ήταν ευτυχείς, αλλά και στο Συμβούλιο. Ε, υπήρξε μεγάλο χάσμα μεταξύ προοδευτικών χωρών και άλλων που δεν ήθελαν να προωθηθεί αυτή η πολιτική, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία δυστυχώς ε, σε επίπεδο Υπουργών Βιομηχανίας και Υπουργείου Μεταφορών. Χαιρόμαστε που προωθεί με αυτές τις πολιτικές και θα ήθελα να πω στην Επιτροπή, ναι, προωθήσατε την πρόταση, αλλά δεν είναι συχνό φαινόμενο το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να καταστήσουν την πρόταση πιο φιλόδοξη. Παλαιότερα η Επιτροπή ήταν ο μεσολαβητής, ε, τώρα όμως υπάρχουν βελτιώσεις και από τις δύο πλευρές ως προς τις κλιματικές αλλαγές. Ως προς τους στόχους χρειάζονται άμεσα έτσι ώστε να υπάρχει καινοτομία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και στην Ευρώπη και βλέπετε ότι ακόμα και η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία μιλά για πλήρη ηλεκτροδότηση των μεταφορών. Βλέπετε λοιπόν ότι και στη Γερμανία προωθούνται τα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλη σημασία ο, η ρύθμιση και ο διακανονισμός. Η κυρία Κόνετσνα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Αν ήθελα απλώς να δω τα αποτελέσματα διαπραγματεύσεων θα μπορούσα να πω ότι είμαι ικανοποιημένη από την έκβαση. Ήταν πολύ καλή η διαδικασία και είμαστε ευγνώμονες ε, προς την κυρία Ντάλη. Όμως ε, υπάρχουν πολλά αιτήματα. Εδώ είμαστε στην απαρχή μιας πορείας. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα νέα καθαρά οχήματα αλλά η πρόταση δεν είναι αρκούντος φιλόδοξη. Έχουμε κάπως καθυστερήσει. Θα ήθελα να πω τι θα κάνουν οι κατασκευαστές, σε ποιους θα απολύσουν αυτοκίνητα, ποιος θα είναι σε θέση να αγοράσει αυτά τα οχήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνει το άγχος στους ε, κατασκευαστές και μόνο. Ε, πρόκειται για την ε, αχιλιοπτέρνα της αγοράς, αλλά κανένας δεν θέλει να εκινήσει αυτή την αγορά, γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα φτάσουμε σε μια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων είναι το πρώτο βήμα, αλλά έχουμε ανοίξει τους ασκούς του αιώλου. Επρόκειτο για ένα πακέτο και δεν έχουμε κάνει αρκετά. Ευχαριστούμε πολύ από το EFTD η κυρία Εύη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το 2017, εξαιτίας της ε, κατανάλωσης ε, πετρελαίου, οι εκπομπές αυξήθηκαν στην Ευρώπη, καθώς και το διοξίδιο του άνθρακα στα νέα οχήματα. Βεβαίως τα αυτοχήματα ντίζελ μειώνονται και τα υβριδικά αυξάνονται. Αλλά το 19 υπάρχουν 20 μόνο τέτοια μοντέλα στις αντιπροσωπίες. Αυτό μας δείχνει ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε αυτό το πλαίσιο για την απομάκρυνση από τον άνθρακα στον ε, τομέα των οχημάτων και των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων έτσι ώστε να φτάσουμε στις μηδενικές εκπομπές. Εγώ είμαι υπερήφανη διότι συνεισέφερα από πλευράς του κινήματος ε, πέντε αστέρων έτσι ώστε να μειωθεί και η χρήση ορυκτών καυσίμων. Αυτό σημαίνει ότι θα επενδύσουμε στις ανανεώσιμες και το υδρογόνο και θα δημιουργήσουμε 200.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2030 έτσι ώστε η μετάβαση να είναι δίκαιη και να μην μείνει κανείς πίσω. Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Ντάλη. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Λαντσίνη για 1,5 λεπτό από το ΕΝΕΦ. E Ευχαριστώ πρόεδρε. Η στόχη μείωσης διοξιδίου του άνθρακα αυτής της πρότασης δεν είναι ρεαλιστική. Δεν λαμβάνουν υπόψη την ε, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, αλλά και τεχνολογική. Γιατί ε, απασχολούνται 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε αυτόν τον τομέα, και εάν μιλάμε για ηλεκτρικά οχήματα, η Ευρώπη δεν θα χρειάζεται πρώτες ύλες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα είναι ε, θα εξαρτάται από την Κίνα για την αγορά συσσωρευτών και δεν υπάρχουν και υποδομές ανατροφοδότησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρησιμοποιούμε μονάδες λιγνίτη για την κατασκευή αυτών των οχημάτων. Γι' αυτό θα πρέπει ο τομέας αυτός να έχει μία μακρόπνοη ε, προοπτική, διαφορετικά είμαστε εντελώς ανεύθυνοι. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λίζε έχει το λόγο για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Η προστασία του κλίματος ε, και η προστασία της απασχόλησης πρέπει να συμβαδίζουν, να πηγαίνουν χέρι με χέρι. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό σε αυτό το νομοθέτημα να δούμε τι επιπτώσεις ε, θα υπάρξουν για την απασχόληση της εργασίας ε, και η Κομισιόν έχει κάνει σοβαρό αντίκτυπο, ε, μελέτη, σοβαρή μελέτη αντικτύπου και είμαι ευγνώμων. Ήταν σαφή λοιπόν τα αποτελέσματα. Υπάρχουν προτάσεις 75% ή 50% αρχική πρόταση ντάλι, αλλά θα είχε αυτό κοστίσει σε θέσεις εργασίας. Η 50 αρχικη προταση νταλι αλλα θα ειχε αυτο κοστισει σε θεση εργασιας η αναλυση της Κομισιόν ε, λέει ε, πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα αντικρούσει. Δεν έχω συναντήσει εγώ τουλάχιστον. Ε, δεν έχω συναντήσει. Δείχνει ανάλυση ότι τελικά είναι λάθος να λέει κανείς ότι όταν είμαστε πάνω από το 30% θα έχουμε καταστροφικές συνέπειες. Αντίθετα, δείχνει η Κομισιόν ότι όταν μείνουμε γύρω στο 40% και νομίζω ότι είμαστε κάτω με ένα περιθώριο ασφάλειας, μπορούμε να έχουμε θετικές επιπτώσεις συνολικά για την απασχόληση στην Ευρώπη. Και δεν θα ήταν ευφυές να μην είχαμε αξιοποιήσει τα περιθώρια αυτά. Όταν δε πολλοί, ιδίω νέοι στην Ευρώπη, ε, περιμένουν από εμάς μέτρα για την προστασία του κλίματος. Είναι λοιπόν μια θετική συμβεβαστική λύση και ελπίζω αύριο ε, με μεγάλη πλειοψηφία να υποστηριχθεί. Όλοι έχουμε συνεισφέρει, βέβαια η συγκίτρια πάνω απ' όλα, αλλά και ο Γιάννης Γκίζη και κυρίως από το ΕΛΚΟ, ο Επίτροπος Μιγγελαρίας και η Ελίζα Μπεθκέστιγκερ από την Προεδρία του Συμβουλίου. Το αποτέλεσμα είναι καλό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρώπη είναι κίνηση. Κίνηση προς νέα μοντέλα ανάπτυξης. Μία οικονομία με μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Μιλάμε για παραγωγή και βιομηχανία με χαμηλότερη μόλυνση. Το 2050 θα έχουμε αύξηση κατά 40% της κινητικότητας των ανθρώπων και 60% των εμπορευμάτων. Ε, δυστυχώς οι μεταφορές είναι υπόλογες για το 25% των εκπομπών και 70% για τις οδικές μεταφορές. Σήμερα οι μεταφορές είναι το 5% του κοινοτικού ΑΕΠ, ε, χωρίς να λάβουμε υπόψη την μόλυνση που οδηγεί και σε κλιματικές αλλαγές. Ο κανονισμός ορίζει δεσμευτικούς κανόνες σε σχέση με τις εκπομπές ιδιαίτερα των ελαφρών οχημάτων. Μιλάμε για ένα τέρμα στις δοκιμές σε συνθήκες εργαστηρίου. Τώρα εργαζόμαστε όλοι για να προωθήσουμε τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις για την μετάβαση και μετατροπή του τομέα, έτσι ώστε να μην εξαρτάται κατά 95% από το πετρέλαιο. Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι θα ε, πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και αυτός ο κανονισμός ε, είναι ένα βήμα προς αυτή την ε, κατεύθυνση υπέρ του περιβάλλοντος. Λούγκρεν, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τα θέματα του περιβάλλοντος απαιτούν από εμά να θέσουμε στόχους. Πριν όμως ρεαλιστικούς. Μόνο έτσι οι κατασκευαστές θα μπορέσουν να υιοθετήσουν νέα τεχνολογία και να μην αποτύχουν. Γιατί η ουσία είναι επίτευξη των στόχων, οι οποίοι πρέπει να είναι όμως στόχοι, όπως είπα, εφικτοί. Ε, εγώ που ζω σε μια αγροτική περιοχή και είμαι ευχαριστημένος από το αυτοκίνητό μου, όμως στις πόλεις που δεν υπάρχουν αρκετά σημεία επαναφόρτησης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τι θα γίνει. Μπορεί να τα καταφέρω στη δική μου περιοχή, αλλά τι θα γίνει αλλού. Εγώ στην περιοχή μου μπορώ να επαναφορτήσω πολύ εύκολα, αλλά ακόμα στις πόλεις αυτό δεν είναι δυνατόν. Ε, δεν είναι λοιπόν εναλλακτική λύση για όλα. Ευχαριστώ. Μπλε κάρτα. Κύριο Ρούμπιχ, ευχαριστώ πολύ. Ε, γιατί ω ε, ε, γίνεται πολλής λόγος ε, και πόσο κοστίζει ή μάλλον πόσα κιλά είναι το με το σχάρι τα 70 αλλά μπορεί κανείς να πάει 700 χιλιόμετρα ενώ με την ηλεκτροκίνητο όχημα 350 άρα υπάρχει θέμα μεγάλης αποδοτικότητας θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας άποψη κύριε Λουγκρή ήταν μπλε κάρτα από τον κύριο Ρούμπιχ ναι, ακούστε κύριε Ρούμπιχε, ακριβώς γι' αυτό το λόγο ε, έχω κι εγώ ένα κανονικό αν θέλετε αυτοκίνητο με κινητήρα καύσης, ε, τα ηλεκτρικά οχήματα πράγματι, μπορεί να καλύψει κάποιες διαδρομές, όχι, δεν είναι όμως κατάλληλο για όλες τις διαδρομές. Διακόπτει ο πρόεδρος. Ε, γιατί κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τη διερμηνία. Μπορείτε να επαναλάβετε κύριε Λούγκριν γιατί δεν μεταφραστήκατε σε όλες τις γλώσσες. Ναι, λοιπόν έλεγα για τα ηλεκτρικά οχήματα ότι δεν μπορεί να λειτουργούν παντού και πάντα. Και εγώ κάνω 70 χιλιόμετρα τη μέρα. Μπορώ να το κάνω με ε, το ηλεκτρικό όχημα, αλλά υπάρχουν προβλήματα, παραδείγματος χάρη το χειμώνα. Μπορεί να καλύψει κανείς πολύ λιγότερα χιλιόμετρα. Υπάρχουν λοιπόν ε, και εναλλακτικέ. Έχουμε και τα κάψιμα, τα φιλοπεριβαλλοντικά, ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Οι ηλεκτρικά οχήματα δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα, αλλά μόνο ένα μέρος των προβλημάτων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι σε δύο-τρία χρόνια που θα τα ξαναλέμε θα θυμούμαστε με νοσταλγία την παλιά τεχνολογία. Ξέρετε, τα πράγματα εξελίσσονται τόσο γρήγορα που εμείς ε, ως νομοθέτες σε κάθε περίπτωση θα βγούμε καθυστερημένοι. Θέλω να πω ότι οδηγούμε τα diesel στο γκρεμό για να δούμε νέα τεχνολογία στους αυτοκινητοδρόμους. Η BMW χθε ανακοίνωσε νέα γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων με αυτονομία 600 χιλιόμετρων και ότι θα επενδύσουν 44 εκατομμύρια στη νέα τεχνολογία τα επόμενα χρόνια. Θα υπερψηφίσω τον συμβασμό ε, αν και ξέρω ότι σε δύο-τρία χρόνια όλα αυτά θα είναι ήδη παροχημένα γιατί η αγορά εξελίσσεται πιο γρήγορα και από εμά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Τελούντε, τον επόμενο μιλητή. Μπόιλεν, παρακαλώ. Πρόεδρε, η κοινωνία των πολιτών μα επεφημεί από πέρσι γιατί υιοθετήσαμε μια σκληρή στάση και υιοθετήσαμε ένα φιλόδοξο όραμα πιέσαμε την βιομηχανία να κάνει αυτό που πρέπει για το περιβάλλον. Αυτό που είναι όμως απογοητευτικό στην τελική συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν είναι ότι οι Υπουργοί είναι τελικά ικανοποιημένοι με μια μερική νομοθεσία η οποία όμως δεν κάνει αρκετά για τη μεγαλύτερη πηγή ρήπαν στον πλανήτη. Οι κουμπές αυξάνονται, δεν βελτιώνεται υπαρκώς γρήγορα η φιλικότητα προς το περιβάλλον των αυτοκινήτων. Χρειαζόμαστε νέες συμφωνίες με πιο αισιόδοξου με πιο απαιτητικού στόχους. Αυτό είναι καθήκον του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου. Όλοι έχουμε να, πρέπει να λάβουμε τις ευθύνε μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μόιτεν έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα μιλάμε για τη σχιζοφρένεια ε, την οποία ε, εκφράζουν ε, στο σώμα αυτό αυτές οι νέες απαιτήσει σε σχέση με τις εκπομπές του άνθρακα από τα βατικά οχήματα. με μεγάλη μανία Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν να βρίσκεσαι σε οικονομία κεντρικού σχεδιασμού προσπαθεί να προωθήσει μια βιομηχανική στρατηγική που ουσιαστικά θα αποτελειώσει το δυνατό χαρτί μας που είναι η αυτοκινητοβιομηχανία. Θέλουμε μηδενικές ε, εκπομπές για να προωθήσουμε την ηλεκτροκίνηση. Από επιστημονική πλευρά αυτό θα οδηγήσει αταξία και από φυσική πλευρά δεν μπορεί να γίνει. Ε, αυτό δείχνει κυρία Ντέλη ότι δεν καταλαβαίνετε γιατί μιλάτε. Από την άλλη πλευρά κάτι άλλο το οποίο συζητούμε εδώ είναι πώς ε, θα βάλουμε στο στόχο τους μεγάλους ε, κατασκευαστές αυτοκινήτων από τη Γερμανία και να αποδυναμώσουμε στη Γερμανία, ξεχνώντας ότι περιμένετε από την άλλη να στηρίξουμε οι Γερμανοί ε, τις τράπεζες, την πολιτική συνοχή, τις επιδοτήσεις, την ανταγωνιστικότητα. Σταματήστε λοιπόν, εγκαταλείψτε αυτή την προσπάθεια και αυτό δεν το λέω μόνο για εσάς, αλλά ισχύει και για μένα και για την γερμανική κυβέρνηση που πάσχει από την ίδια χιζοφρένη ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκούτελαντ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Σουηδία είναι μία από εκείνες τις χώρες όπου ε, βασιζόμαστε στην αυτοκινητοβιομηχανία. Θέλουμε να προωθηθούν οι κατάλληλοι όροι για μια βιώσιμη βιομηχανία για την επαύριον. Γι' αυτό οι σοσιαλδημοκράτες και εδώ αλλά και στην πατρίδα μας προσπαθήσαμε να ορίσουμε τους στόχους υπέρ του κλίματος και του περιβάλλοντος γιατί θέλουμε μείωση των εκπομπών ε, ακόμα περισσότερες από αυτές που βλέπουμε σε αυτό το κείμενο. Αλλά ε, η δική μας εισηγήτρια η Μίρια Μτάλη κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έχουμε νέους κανόνες υπέρ του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες αύριο θα ταχθούμε υπέρ της δημόσιας υγείας του περιβάλλοντος και μίας αυτοκινητοβιομηχανίας που θα κατέχει ε, μία εύρωστη θέση για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Κέλμελ, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ ε, μακριά από την πραγματικότητα αυτό το σχέδιο εξ ό,τι αφορά στους στόχους ε, και ουσιαστικά είναι πάλι ιδεολογικό το ζήτημα. Ε, και η ιδεολογία που επικρατεί δείχνει ότι ουσιαστικά είμαστε κατά τη ιδιωτική κινητικότητα. Ακούσαμε διάφορα επιχειρήματα που δεν ευσταθούν καθόλου. Και ο Επίτροπο Κανιέται λέει ότι θέλει αυτοκίνητα που δεν εκπέμπουν καυσαέρια. Αυτό είναι ουτοπία γιατί δεν υπάρχει ε, δυνατότητα μηδενικών εκπομπών. Ούτε προβλέπεται στο μέλλον να το πετύχουμε. Και μιλάμε για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Υποτίθεται ότι αυτά θα φέρουν τη σωτηρία αυτά είναι νοησίες ε, κυρίες και κύριοι, γιατί καταναλώνουν ρεύμα. Και από πώς, ε, θα παράγεται αυτό το ρεύμα στα θερμελεκτρικά εργοστάσια στη Γερμανία ή ε, με, και έχοντας πετρέλαιο θα είναι λοιπόν ουτοπικό ότι θα προκύψει τόσο μεγάλη βελτίωση. Ε, το ηλεκτροκίνητο όχημα για να κυκλοφορήσει θα έχει μολύν το περιβάλλον ε, πάρα πολύ ε, περισσότερο, το ίδιο τουλάχιστον με τα άλλα οχήματα, τα οποία μπορεί να κάνουν και πολύ μεγάλες αποστάσεις και μην μιλάμε και μην αφήνουμε εκτός, μιλώντας μόνο για τις οδικές μεταφορές, την αυτιλία. Γιατί τα μεγάλα πλοία, τι ακριβώς το ίδιο και να μην πω και περισσότερο, πολύ περισσότερο το μολύνουν το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αυτός ο κανονισμός μας δίνει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για να φτάσουμε στους στόχους της συνθήκης του Παρισιού τα επόμενα χρόνια με την σύσταση αυτών των στόχων έχουμε ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό για τις επενδύσεις και την τεχνολογική εξέλιξη. Ο τομέας του ε, τουρισμού έχει μεγάλη σημασία για πολλές χώρες όπως η δική μου και τα κράτη-μέλη θα ε, γνωρίσουν μία μεγάλη αλλαγή και μετασχηματισμό. Αλλά αυτή η μετάβαση σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι στόχοι του περιβάλλοντος τη στιγμή που αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα. Και γι' αυτό θα πρέπει να επαγρυπνούμε σε επίπεδο περιφερειών και τοπικών αρχών που είναι πιο ευάλωτες, διότι εδώ δεν μιλάμε ε, μόνο για την αυτοκίνητο βιομηχανία, αλλά και την βιομηχανία εξαρτημάτων. Και γι' αυτό θα πρέπει να προβούμε σε αναλύσεις και ειδικά μέτρα για τους πιο σημαντικούς βιομηχανικούς τομείς. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τα επερχόμενα ε, χρόνια, θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ κύριε Επίτροπε για την εξαιρετική εργασία κατά τη θητεία αυτή και γιατί έχουμε πλέον έναν οδικό χάρτη ενώπιον των ευρωεκλογών καθώς και μια στρατηγική για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Ευχαριστώ κύριε Ζρούμπη και έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. 44 δις ε, ε, επενδύσεων ε, λέμε ε, ότι γίνονται. Ουσιαστικά θα είναι πολύ πιο ε, δαπανηρά τα αυτοκίνητα στο μέλλον, άρα είναι και κοινωνικό το ζήτημα για, πολλούς, ε, για πολλά κράτη. Κάποιοι συμπολίτε μας αρκετοί δεν θα μπορούν πλέον να αγοράσουν αυτοκίνητο. Ένα πρόβλημα αυτό. Δεύτερον, μετράμε τα καυσαέρια. Αλλά υπάρχει το ζήτημα της παραγωγής και της ανακύκλωσης και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Για το ντίζελ άλλα. Ε, λέμε ότι ε, η βενζίνη ουσιαστικά ε, εκλεί τα περισσότερα γραμμάρια από καυσαέρια και το ντίζελ τα λιγότερα, 19 περίπου. Θα πρέπει όμως να περάσουμε στην ε, κατάργηση της ε, ατομικής ενέργειας γιατί είναι πάρα πολύ κακή για το περιβάλλον. Πώς θα εξασφαλίσουμε την ε, ηλεκτροκίνηση για όλα αυτά τα οχήματα. Σάλτε Εάν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να φτάσουμε στους στόχους του Παρισιού μετά το 2050 με χαμηλές εκπομπές, τότε το μέα των μεταφορών θα πρέπει να συνδράμει. Γι' αυτό κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση με αυτό το νομοθέτημα. Γιατί γιατί τα οχήματά μας θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον με χαμηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων προς την Μίριαν Ντάλι που προώθησε αυτό το κείμενο μέσα σε μια επίπονη πορεία. Θα μπορούσαμε βεβαίως να έχουμε μείωση 45% ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, δηλαδή να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε νέους που επιμένουν να είμαστε πιο φιλικοί προς το περιβάλλον. Δεν φτάσαμε όμως σε αυτό τον στόχο. Ε, ε, δεν ε, οφείλεται το σφάλμα σε μας, αλλά στο Συμβούλιο. Ο τομέας των μεταφορών θα πρέπει να συνδράμει στους στόχους υπέρ του κλίματος. Εγώ θα υποστηρίξω αυτό το νομοθέτημα γιατί είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει το Συμβούλιο να το ελέγχουμε άμεσα έτσι ώστε να συνδράμει και να αποδώσει. Γκάμπους. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ντάλη καθώς και τον κύριο Χίσεκε για τις διαπραγματεύσεις για να φτάσουμε σε αυτή την έκθεση. Αυτό σημαίνει μεγάλη συνδρομή για την απομάκρυνση από τον άνθρακα και να φτάσουμε σε μια σωστή μετάβαση για την τεχνολογική ουδετερότητα η έκθεση που θα ψηφίσουμε αύριο αφορά μια επίπονη εργασία για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών κατά την θητεία του Προέδρου Γιούνκερ και με τη συνδρομή του Αρίας Κανιέτε. Εμείς θα θέλαμε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Πρόκειται για έναν αγώνα και μία μάχη που δεν μπορούμε να χάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Ζωρίνιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμούμε αυτή την ενεργειακή μετάβαση για τα νέα οχήματα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Μιλάμε για καινοτομία με νέες τεχνολογίες και μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έτσι πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξουν απάτες σαν αυτές που είδαμε στην περίπτωση του Dieselgate. Γι' αυτό χαιρετίζω την εργασία της ε, εισηγήτριας Μίριαμ Ντάλι για αυτή την ισορροπημένη πρόταση που μας επιτρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία καθώς και να προωθήσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη την οποία θα πρέπει να ελέγξουμε και να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους σε όλες τις περιφέρειες υπέρ της καινοτομίας. Ευχαριστώ κύριο Σμιτ. Η κυρία Σμιτ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε την γενική εικόνα. 3% των ετησίων εκπομπών είναι ανθρωπογενείς. Από αυτά 9% είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτό 30% είναι οι συγκοινωνίες και από αυτό πάλι 72% ε, οι οδικές και από αυτό πάλι ένα 60% τα οχήματα που καλύπτει αυτή η πρόταση. Δηλαδή μιλάμε για 0,031% εξοικονόμηση το πολύ. Για ποιον λοιπόν ε, φτιάχνουμε αυτά τα ακριβά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και βλάπτουμε την βιομηχανία μας. Είναι τελείως δυσανάλογα αυτά τα μέτρα. Ειδικά εάν μετρήσουμε μόνο το τι γίνεται στην εξάτμιση, ακόμα και αν το ρεύμα παράγεται από ε, άνθρακα. Βεβαίω, μια πράσινη πλειοψηφία εδώ πέρα και αριστερή θέλει αυτές τις αλλαγές. Μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα και για τους πολίτες μας και για το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπλάνκο Λόπες, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάθε νέα έκθεση που εξετάζουμε μας φέρει ενώπιον της πραγματικότητας και της επιτακτικής ανάγκης να αντιμετωπίσουμε με πυγμή και αποφασιστικότητα τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και που είναι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Σίγουρα οι μεταφορέ είναι υπεύθυνε για το 1 τέταρτο των εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε η απαλλαγή μα από εκπομπέ άνθρακα στι μεταφορέ είναι υποχρέωση και όχι επιλογή η προαίρεση. Σίγουρα ο συγκεκριμένο κανονισμό μα βάζει στο μονοπάτι για να υλοποιήσουμε αυτού του στόχου και να απαλλαγούμε από εκπομπέ άνθρακα. Είναι αναπόφευκτο αυτό ο στόχος. Επίση, ε, αντιμετωπίζουμε την πρόκληση να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα